Okay, colleagues, we can now make a start. We're waiting for... Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Περιμένουμε τον εισηγητή για την πρώτη ψηφοφορία. Θα ήθελα καταρχήν να πω στους συντονιστές ότι είχαμε σκεφτεί η συνεδρία να προχωρήσει μετά την ψηφοφορία κατευθείαν, αλλά κάποιοι συνάδελφοι είχαν πρόβλημα με αυτό, οπότε 11.30 11 ε, θα, έρθουν οι συντονιστές. Ήταν περίπλοκο ιδάλλως να αλλάξουν τα σχέδια. Οπότε, στις 11.30 οι συντονιστές, στη συνέχεια ε, να θυμίσω στις 3 η ώρα έχουμε μια συνάντηση και στις 5.30 επίσης όπου θα μιλήσουμε για DG Echo Λοιπόν, ήρθε ο Ιγνάθιο, οπότε θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία με την ε, έκθεση, το σχέδιο έκθεσης για την πρόσβαση στα φόρμακα. Ιγνάθιο, θες να πεις κάτι πριν ξεκινήσουμε. Όχι, πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία λοιπόν. Να κάνουμε ένα τεστ πρώτα, μια δοκιμή. Λοιπόν, άρτη ψηφοφορία. Δοκιμαστικά, έτσι. Κάποιος δεν έχει ψηφίσει. Εντάξει, ναι, λειτουργεί. Πολύ ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Με το συμβαστικό α, συμβαστικό κείμενο α, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Β, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Όλες οι... Προφορική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ναι, το 9 να το ε, ελέγξουμε παρακαλώ. Άρχιτη ψηφοφορία. Α, είναι σαφέστερα τώρα τα πράγματα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός Γ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ τροπολογία 25 άρχιτη ψηφοφορία τώρα είναι σαφέστερα τα πράγματα πέρας ψηφοφορίας ναι, απλώς είδα διαφορετικές ενδείξεις προηγουμένως. Τροπολογία D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λοιπόν, ε, συμβασμός ε, δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην 49, τροπολογία 49, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές το ελέγξουμε παρακαλώ 53 άρχιτη ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 54 υπέρ Κατά αποχές απορρίπτεται. 55. Α, σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος 55. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος της 55. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο μέρος τώρα του 55, έχει τρία μέρη 55, συγγνώμη. Ναι, τρίτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 56, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59, υπέρ, κατά αποχές να το ελέγξουμε το 59 παρακαλώ άχτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται G τώρα ε, συμβασμός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβασμός F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα στο 72. Τροπολογία 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός H. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 77, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78, σε δύο μέρη, 78. Πρώτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε το πρώτο μέρος του 78. Παρακαλώ, άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος. μέρο. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του συνόλου νομοδότησης άρχιτη ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας και τώρα βλέπω ότι είναι μεγάλη πλειοψηφία Συγχαρητήρια Ιγνάθιο και συγχαρητήρια και για τη δουλειά σας στους συμβασμούς ε, διότι έτσι είναι πιο απλή και ψηφοφορία και είναι και πιο σαφές το μήνυμα τελικά. Λοιπόν, και τώρα να περάσουμε στην πρώτη ε, του κυρίου Πέντα. Έχουμε δύο εκθέσεις. Η πρώτη είναι μια σημαντική έκθεση του Christian Van για την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας στον τομέα της ανάπτυξης. Ωραία, να ξεκινήσουμε με το συμβασμό 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε. Τροπολογία 55 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται οριακά. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 4. Εδώ τα ψηφίζουμε όλα μαζί. Τους ε, συμβασμούς 4 έως 7 αν δεν έχετε αντίρρηση. Λοιπόν, 4 έως 7. Ποιοι είναι υπέρ. Συμβασμοί 4 έως 7. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε. Έχουμε τώρα τον συμβασμό τον, την τροπολογία 62, συγγνώμη, τροπολογία 62 υπέρ. Κατά αποχές να το ελέγξουμε. Παρακαλώ τροπολογία 62, άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές ξανά 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 83 παρακαλώ άρχιτε ψηφοφορία για την 83 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές 86 παρακαλώ οι συντονιστές σας μας πούνε είναι πιο εύκολο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την τροπολογία 87 παρακαλώ άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας Εγκρίνεται η 87. Το 6 το κάναμε. Το στο... Λοιπόν, τροπολογία 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε την τροπολογία 99 παρακαλώ. Άχτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα συνολικά ψηφίζουμε για τους συμβασμούς 9 έως 12. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 108. Υπέρ, κατά, αποχές 108 ξανά υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την τροπολογία 108 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 να ελέγξουμε 118 ελέγχουμε άρχιτη ψηφοφορία μου φάνηκε σαφές αλλά ας το ελέγξουμε πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται είχατε δίκιο να δείχνετε παρακαλώ ότι ψηφίζετε 119 119. 119 δεκαεννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα... Όχι, αυτό το κάναμε. 123 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε 123 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την τροπολογία 6 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε από κοινού του συμβασμού 13-17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την τροπολογία 12 άρχισε ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε το 15. η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε την τροπολογία 18 παρακαλώ. η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές να απορρίπτεται 32 υπέρ κατά απορρίπτεται 33 υπέρ όχι 33 το κάναμε συγγνώμη 33 είναι 33, 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ δεν μπορείτε να ζητήσετε έλεγχο άμα εθνίστε βουλευτής. 34 ε, λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Όχι 35. Όχι 36. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 ε, συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα <clears throat> για το 10 εδώ τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί του συνόλου. Άρχιτη ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Πρέντα για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Πολύ καλή συνεργασία. Ε, Πήγαμε πολύ καλά και στην ψηφοφορία. Okay, we can move to the next item, which is... Περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση για την προώθηση ισότητας φύλων στην ψυχική υγεία και κλινική έρευνα. Ο Φλωρέντ Μαρτσελέζη είναι εισηγητής. Θα ψηφίσουμε για τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές. Σας παρακαλώ να βλέπω καλύτερα υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε την ε, τροπολογία υπαριθμών 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε συμβαστική α. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία βλέπετε. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Τροπολογία 10. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση στο σύνολό της. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία να συγχαρούμε τον εισηγητή. Ο κύριος Γκερέιρο θέλει το λόγο. Απλώς θα ήθελα ε, να συγχαρεί η Επιτροπή των Ζόρντι Σεμπαστιά για την έκθεση αυτή γιατί δεν είναι μέλος του Κοινοβουλίου, έχει αντικατασταθεί, αλλά έτσι αναγνωρίζουμε την εργασία του. Ναι, αυτό μπορεί να μπει στα πρακτικά. Ο κύριος Σεμπαστιά αποχώρησε από το Κοινοβούλιο και έχει αντικατασταθεί, άρα θα πρέπει να τιμήσουμε την εργασία του και να τον ευχαριστήσουμε για την ε, γνωμοδότηση αυτή. Σας ευχαριστώ κύριε Γκερέιρο. Βλέπουμε ακόμα και από αντίπαλα κόμματα υπάρχει αναγνώριση της εργασίας. Λοιπόν, προχωρούμε στην ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΚΤΟ. Ο κύριος Λούκε είναι εισηγητής. Θέλετε κάτι να πείτε? Όχι, ωραία, περνάμε στην ψηφοφορία. Συμβαστική Β, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Γ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. 15 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Συμβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 22 υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της 22. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πράγματι. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όχι, όχι, ελέγχουμε την 26. Άρχεται η ψηφοφορία για την 26. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται με πολλές αποχές. 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. F υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 36 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε στο σχέδιο γνωμοδότηση, στο σύνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Και εγώ βέβαια. Εμείς συμπεριλαμβανομένης. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία να συγχαρούμε τον κύριο Λούκε. Σας ευχαριστούμε πολύ ιδιαίτερα για τις συμβιβαστικές γιατί έτσι πέρασε και γρηγορότερα, εγκρίθηκε γρηγορότερα η έκθεση. Τώρα, περνάμε στην επόμενη έκθεση του κυρίου Πρέντα. Είναι γνωμοδότηση για την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο για το 2015. Κύριε Πρέντα, θέλετε κάτι να πείτε. Ωραία. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε τη 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται πρέπει να ψηφίζετε με σαφήνεια. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές ε, παρακαλώ να ελέγξουμε την 20 ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της 53 υπέρ κατά Αποχές ελέγχουμε το πρώτο τμήμα της 53, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της 53 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε την 54, αρχίζει η ψηφοφορία 54 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ελέγχουμε την 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε 71 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73. Θέλουμε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 72. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Είχατε δίκιο. Είχατε δίκιο. Ε, δυστυχώς φαίνονται τα χέρια πολύ αργά. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ναι, ναι, απορρίπτεται. Με μεγάλη πλειοψηφία. Ε, 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίσουμε στο σχέδιο της γνωμοδότησης, στο σύνολό του, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Να συγχαρούμε και πάλι τον κύριο Πρέντα. Τώρα έχουμε την τελική ψηφοφορία σε σχέση με την πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έκθεση της κυρίας Μακάβαν. Συμβαστική 1. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά. Διακόπτη πρόεδρος. Μια στιγμή παρακαλώ. Είμαστε στην προφορική ερώτηση. Έχετε δίκιο κύριε Πρέντα δεν το είχα στι σημειώσει. Πρώτα έχουμε την προφορική ερώτηση, έχετε δίκιο, και μετά έρχεται το ψήφισμα. Ξαναρχίζουμε λοιπόν με την προφορική ερώτηση, τι οποίε δεν υπάρχουν τροπολογίε. Θα κάνουμε λοιπόν μια ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία για την προφορική ερώτηση. Πάλι καλά, το Λαϊκό Κόμμα είναι ξύπνιο σήμερα και μας βοηθεί. Ψηφίσατε όλοι και όλες ε, λίγοι. Εγκρίνεται λοιπόν η προφορική ερώτηση και με μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε το ψήφισμα. Ξαναρχόμαστε λοιπόν στο ψήφισμα για την πρόσβαση στην ενέργεια σε αναπτυσσόμενες χώρες. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. 69, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συν Τροπολογία 70 υπέρ. Κατά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 εδώ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Πρώτο τμήμα της 78 αρχίζει. Πέρας, απερίφθη. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορριπτωτική και αυτό. 79 υπέρ, κατά, αποχές επαλήθευση αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε πέρας εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 Α, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της 81 υπέρ. Κατά. Αποχές επαλήθευση για το πρώτο τμήμα της 81. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 81. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 82. Σε δύο τμήματα πάλι. Πρώτο τμήμα της 82. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 82 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση 83 πέρας εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση 85 αρχίζει η ψηφοφορία νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά ίσως και όχι πέρας εγκρίνεται τελικώς 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ. Υπέρ λέω πάλι. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση, επαλήθευση. 89. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έχουμε μόνο το δεύτερο τμήμα της 90 ως προσθήκη. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. ...96 υπέρ... ...κατά... ...αποχές απορρίπτεται... ...97 υπέρ... ...κατά... ...αποχές απορρίπτεται... ...102 υπέρ κατά, αποχές. Θα χρειαστεί επαλήθευση διότι ορισμένες ομάδες δεν ψηφίζεται καθόλου. 102 λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Και απεριφθεί. Δώστε και ένα σήμα κάποιος στις ομάδες. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά αποχές, επαλήθευση, 99, ε, επαλήθευση 99, αρχίζει. Ψεφίσατε όλοι, τέλος, απερίφθη. 98, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθεται. 100, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές να κάνουμε επαλήθευση για την 106 ε, επαλήθευση λοιπόν αρχίζει η ψηφοφορία τέλος απερίφθη 105 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται, ας την επαληθεύσουμε, 105, πέρας, εγκρίνεται. Τώρα τα εκτιμώντα τα citations υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία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 αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση 19 λέει η πρόεδρος αλλά είναι 20 20, 20 διορθώνει αρχίζει ψηφίσατε όλοι πέρας και απερίφθη. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση 33 αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε πέρας εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές Επαλήθευση. Επαλήθευση 35. Δεν σηκώνουν όλοι καθαρά τα χέρια. Πέρας. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση γιατί είναι 36. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ακολουθεί η υπαριθμόν 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή. 44 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. 44 αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. 48 αρχίζει. Ψηφίσατε άπαντες. Πέρας. Απερίφθη. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας την επαληθεύσουμε. Αρχίζει. Πέρας εγκρίνεται με διαφορά τριών ψήφων. 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά αποχές. Επαλήθευση 56. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. Απερίφθη. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση 57. Αρχίζει. Πέρας. Απερίφθη. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε το ψήφισμα στο σύνολό του. Όχι ονομαστικά. Όχι ονομαστικά. Α, ηλεκτρονικά όμως. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Ωραία. Εδώ ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Διάδημα για τους συντονιστές μέχρι τις 11.30.